Dear κάνω κάνουμε μια δοκιμή, αγαπητοί συνάδελφοι. Ψηφίζουμε δοκιμαστικά, ηλεκτρονικά. Έχουμε έναν από το ΕΛΚ παραπάνω από ό,τι πρέπει, Ευρωβουλευτή. Εντάξει είμαστε τώρα. Υπάρχουν ε, συνάδελφοι που δεν έχουν την κάρτα τους και που θέλουν να, μετρηθεί, να μετρήσει η ψήφος τους. Όχι, όλοι, όλοι έχουν τις κάρτες τους, αλλά έχουμε ένα παραπανίσιο από το ΕΛΚ. Ακόμα το ίδιο. Ας το διορθώσουν οι συντονιστές παρακαλώ. Okay.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 μου ζήτησε να ψηφίσουμε την έκθεση του κυρίου Μπαγιέ και της κυρίας Ρέγνερ. Θα ξεκινήσουμε με την τροπολογία 35. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Το θα το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Yes, Υιοθετείτε. Τροπολογία 36 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 37 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 109 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 110 υπέρ κατά άποχες νομίζω ότι απορρίπτεται αλλά θα το ελέγξουμε πέρας ψηφοφορίας Όντως απορρίπτεται. Συμβαστική A, υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετείται. Συμβαστική τροπολογία B, υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετείται. Τροπολογία 131, υπέρ, κατά, αποχές, Απορρίπτεται. Τροπολογία 15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 161 υπέρ. Κατά. Την ελέγχουμε ηλεκτρονικά την 161. έχουμε υπερβολικά πολλούς ευρωβουλευτές από το ΕΛΚ. Δύο παραπάνω για την ακρίβεια. Εντάξει τώρα. Υιοθετείτε. 162 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 163 υπέρ. Κατά. Αποχές. Το ελέγχουμε ε, ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την 163. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 164 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 165 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Λοιπόν, την ελέγχουμε ηλεκτρονικά, 165. Ψήφισμα τώρα. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Okay. Okay. Um, Συμβασμός. Συμβαστική 6. Υπέρ, κατά, αποχές. Υιοθετείτε. Τροπολογία 206 υπέρ. Υπέρ, κατά, αποχές. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά 206. Είναι συμβατή η 206 με την συμβαστική τροπολογία. Ψηφίζουμε τώρα. Έχουμε έναν παραπάνω σοσιαλιστή. Πέρας ψηφοφορίας. Υιοθετείτε. 207 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ελέγχουμε χρονικά 207. ψηφίσουμε τώρα. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται συμβαστική D. Κύριε Ρωσάτη. Πρόεδρε. Ένα διαδικαστικό θέλω να θέσω. Έχουμε δύο εναλλακτικέ συμβαστικές τροπολογίες. Την D που υποβλήθηκε από τους και μία άλλη εναλλακτική ως προ αυτή που υποβλήθηκε από τρεις πολιτικές ομάδες. Με βάση τους κανόνες θα πρέπει να ψηφίσουμε αυτές τις συμβαστικές τροπολογίες. Γιατί αποκλίνουν από το αρχικό κείμενο. Κατά την άποψή μας, η συμβαστική τροπολογία του ΑΛΔΕ είναι πολύ πιο, πάει πολύ πιο μακριά σε σχέση με το αρχικό κείμενο. Σε σχέ... Καταρχάς, σε ό,τι αφορά το χρονικό όριο για την ε, ασφαλιστική ρήτρα, δίνει ένα αόριστο χρονικό διάστημα, ενώ ο συμβιβασμό των συνεισηγητών προσφέρει ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για την εξαίρεση. Και το δεύτερο, για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η συμβαστική του Άλντε πάει πολύ πιο μακριά. Δηλαδή δίνει πολύ περισσότερε εξουσίες στην Κομισιόν. Για αυτό το λόγο προτείνω, Πρόεδρε, να ψηφίσουμε πρώτα την συμβαστική τροπολογία του Άλντε, των φιλελεύθερων. Εύελιν Ρέγνερ. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ δεν συμφωνώ. Συμφωνώ με τον ε, κανονισμό. Οι συμβιβαστικές τροπολογίες θα πρέπει να ψηφίζονται με την σειρά. Ναι, επαναλαμβάνω, βάλτε τα ακουστικά σας. Αλλιώς να μιλήσω αγγλικά. Δεν έχω πρόβλημα. Λοιπόν, εγώ διαφωνώ με αυτή την προσέγγιση. Σύμφωνα με τον κανονισμό θα πρέπει οπωσδήποτε πρώτα να ψηφίσουμε αυτήν τη συγκεκριμένη τροπολογία. Εάν υπάρξουν αμφιβολίες ή επιφυλάξεις, ε, μπορούμε να επικαλεστούμε και τη γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας. Το συζήτησα με τον συμπρόεδρο. Είναι δύσκολη η κατάσταση, γιατί διαφωνούμε μεταξύ μας. Εγώ συμφωνώ με τις δικές μας υπηρεσίες που θεωρούν ότι η συμβαστική τροπολογία D πρέπει να ψηφιστεί πρώτα, γιατί αποκλίνει περισσότερο από το κείμενο της ε, Κομισιόν. Για το λόγο ότι καλύπτει και τις τρίτες χώρες, που είναι η βασική αλλαγή που ρυθμίζει το κείμενο του Κοινοβουλίου. Η συμβαστική D καλύπτει τις τρίτες χώρες. Θα έχουμε λιγότερες εξαιρέσεις από ό,τι με την άλλη ε, τροπολογία. Δηλαδή, με, το, με τη συμβαστική D δεν υπάρχει αόριστη εξαίρεση, ενώ αλλιώς έχουμε εξαίρεση για δύο χρόνια συν δύο. Για τις εταιρείε που τις αφορά αυτή η συμβαστική, με την συμβαστική D, ε, αποκλίνουμε περισσότερο από την ε, πρόταση της Κομισιόν, ενώ με την αναλλακτική είμαστε πιο κοντά στην πρόταση της Κομισιόν, γιατί ε, σας εξήγησα. Κατά την άποψη λοιπόν τη δική μου και Τη υπηρεσία θα πρέπει να ψηφιστεί η συμβαστική D πρώτα. Λυπάμαι που πρέπει να ψηφίσουμε. Έτσι. Εκτός και αν, έχω πείσει το συμπρόεδρό μου, αν και δεν νομίζω. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να αφήσουμε τώρα τα τεχνικά θέματα στην πάντα και να ψηφίσουμε πολιτικά. γιατί ε, υποβάλλουμε τα δικαιώματα μειοψηφίας ε, στην ψήφο της ε, πλειοψηφίας. Επιμένω, κύριε Σβόποντα, να δεχτούμε την ερμηνεία της ε, υπηρεσίας μας, που είναι μια τεχνική ε, ερμηνεία και όχι πολιτική. Ε, Δεν θέλω να παρατείνω τη συζήτηση. Ναι, συμφωνώ με τον κύριο Γκουαλτιέρη ότι πρέπει να ψηφίσουμε πρώτα τη συμβαστική D και την D2 εν συνεχεία, την αλλακτική D μετά. Λοιπόν, εάν δεν θέλετε μυστική ψηφοφορία, να κάνουμε αυτό που είπα. Ε, να ψηφίσουμε δημόσια. Πράσινο πλάς και κόκκινο είναι η εναλλακτική πρόταση του κυρίου Ροζάτη. Το ΣΥΝ είναι η ψήφος που προβλέπεται στην, στον κατάλογο. Ε, το μείον είναι το αντίστροφο. Διαφωνούμε, όπως καταλάβατε, ε, και συμφωνούμε να ψηφίσουμε απλώς. Τι θα ψηφίσουμε τελικά. Εγώ λυπάμαι, γιατί θα έπρεπε να ακολουθήσουμε αυτό που μας είπε η υπηρεσία μας. Λοιπόν, ζητάει κανένα να ψηφίσουμε μυστικά. Όχι, να ψηφίσουμε δημόσια. Ψηφίζουμε λοιπόν τώρα. We Κρατάμε την αρχική δια, ε, σειρά με την οποία θα ψηφίσουμε τις τροπολογίες. Συμβαστική D, λοιπόν. Υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Πέρας Απορρίπτεται. Πάμε την, να ψηφίσουμε την αλλακτική D. Υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά την αναλλακτική D. It Άρα, πάμε στη 221. 221. Υπέρ. Κατά. Την ελέγχουμε χρονικά. Πέρας φοφορίας Απορρίπτεται. ...230 υπέρ... ...κατά... ...αποχές... ...απορρίπτεται... ...231 υπέρ... ...κατά... Α, ...ελέγχουμε τη 231... ...ηλεκτρονικά... ...ψηφίζουμε τώρα... Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 2.32 υπέρ. Κατά. Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά το ελέγχουμε γιατί είδα πολλά χέρια σηκωμένα. Λοιπόν, ψηφίζουμε χρονικά τώρα τη 232. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβαστική Ή. E. Υπέρ. Κατά. Αποχές υιοθετείται. 236 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 237 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχω. Ελέγχουμε χρονικά τη 237. Πέρας φοφορίας. Απορρίπτεται. 238 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 239 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 240 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 241 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Ψηφίζουμε τη 241 και 242 που είναι ίδιες. Πέρας φοφορίας απορρίφθηκαν. 2.43 υπέρ κατά, αποχές υιοθετείται 2.44 υπέρ, κατά. Την ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Πέρας φορείας απορρίφθηκε. 2.45 και 31 και 28. 2.45, 31, 28. Κατά αποχές απορρίφθηκε. 2.46 και 2.47 και 2.48. Όχι, συγγνώμη. Οι 2.46 και οι 2.47 μόνο. Υπέρ, κατά, άποχες. Υιοθετούνται. Ελέγχουμε τη 246 και 247 ηλεκτρονικά. Πέρες απορρίφθηκαν. Πού ήμουν? 248 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. Ελέγχουμε τη 248, αφού το θέλετε. Ψηφίζουμε τώρα. Πέρας φοφορίας. Απορρίφθηκε. 249 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Όχι, δεν θα το ελέγξω. Ήταν προφανές. 259 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 260. Δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα. Οκ, το ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Το πρώτο τμήμα, έτσι. Υιοθετείτε. Συγγνώμη. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 261. Ελέγχουμε το δεύτερο τμήμα, 260. Υιοθετήθηκε. Συγγνώμη, να σηκώνω τα χέρια σας. Δεν φταίω εγώ. 261 υπέρ. Κατά. Παρακαλώ ακόμα μία φορά. 261 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 262 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 263 υπέρ. Κατά. Αποχές. Την ελέγχω ηλεκτρονικά. Πέρας φορείας Απορρίφθηκε. Συμβαστική τροπολογία ΕΦΑ Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. Τροπολογία 34 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 266 υπέρ. Όχι, συγγνώμη, 267 υπέρ. Κατά. Ελέγχω ηλεκτρονικά την 267. Πέρας ψηφοφορίας. Υιοθετείτε. Συμβαστική τροπολογία G υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. Πού πάμε τώρα. «271 και 272 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτονται. 38 υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε την 38 ε, ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε τώρα. Έχουμε έναν ε, από το άλλο παραπάνω. Πέρας η Υιοθετείτε με μία ψήφο παραπάνω. Ένα. Υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε την τροπολογία υπαριθμών 1 ε, ηλεκτρονικά τώρα. Λάθος, δεν έπρεπε να την ψηφίσουμε. Έπρεπε να πάμε κατευθείαν στην 39 μετά την υιοθέτηση της 38. Πάμε να ψηφίσουμε 39 υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε χρονικά 39. Sorry. A lot of people to vote, please. Πολλοί ψηφίζουν. Πολλοί. Πέρας προφορίας. Υιοθετείτε. 40 υπέρ κατά άποχες νομίζω ότι υιοθετείται 41 υπέρ κατά ελέγχουμε ηλεκτρονικά τη 41 τώρα ψηφίζουμε τώρα Vote is closed. Πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται με δύο ψήφους διαφορά. 42 υπέρ. Κατά. Κατά. Αποχές. Δεν βλέπω ότι ψηφίζει το ΕΛΚ. Πάση περιπτώσει εγκρίνεται. 45 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 46 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 47 υπέρ. Κατά. Αποχές Ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ε, 47 ηλεκτρονική. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. 48 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. 49 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 50 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 51 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 52 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 53 υπέρ Κατά. Ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά την 53. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας ψηφορίας. Εγκρίνεται. Άρα... Υπάρχει ένα πρόβλημα στο κατάλογο ψηφοφορία που έχω, δεν έχει λογική. Ψηφίζουμε την 55 υπέρ. 55 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Α ελέγξουμε ηλεκτρονικά 55, ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα ψηφορία εγκρίνεται. 58 υπέρ, κατά, ε, ας ελέγξουμε ε, ηλεκτρονικά τη 58 παρακαλώ. Πέρα ψηφορία απορρίπτεται. 56 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται 57 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 59 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 60 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 61 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 62 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 63 υπέρ κατά αποχές ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά ψηφίστε παρακαλώ νόμιζα απορρίφθηκε αλλά ας δούμε πέρας ψηφοφορίας η 63 εγκρίνεται ωραία καλά που ελέγξαμε 64 υπέρ κατά Ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά. 64. Ψηφίστε παρακαλώ. One EPP too many. Ένας επιπλέον ε, ε, ευρωβουλευτής του ΕΛΚ. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβαστική H υπέρ, κατά αποχές. Εγκρίνεται. 65 υπέρ, κατά αποχές. Εγκρίνεται. 75 ε, κατά ε, νομίζω ε, απορρίπτεται αλλά σε ελέγξουμε 75 ψηφίστε παρακαλώ πέρας ψηφορίας απορρίπτεται με μία ψηφοδιο φορά συνδυαστική I υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 80 υπέρ κατά απορρίπτεται. α ελέγξουμε για να είμαστε σίγουροι. Ψηφίστε για την 80 ηλεκτρονικά παρακαλώ. Vote is close. Απορρίπτεται. Με ισοψηφία μάλιστα. 82 υπέρ. Κατά. Αποχή. Ας ελέγξουμε. 82. Ε, Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Με μία ψηφοδιαφορά 81. Ε, Κατά. Αποχές. Νομίζω απορρίφθηκε. Σε ελέγξουμε. Πέρας ψηφοφορίας. Ισοψηφία, μάλιστα. Απορρίπτεται. 82 υπέρ, κατά, αποχές, Συμβαστική J υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική K υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. DV4 υπέρ, κατά, αποχές. Θα ελέγξουμε για την DV4, ψηφίστε παρακαλώ yes. Για την Deve 4, Deve 4. Πέρασε ψηφοφορία. Πάλι σου ψηφία, απορρίπτεται. 96 υπέρ, κατά, αποχές, ε, απορρίπτεται. 5 υπέρ, κατά. Ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά, παρακαλώ, ψηφίστε παρακαλώ. Πέρασε ψηφοφορία. Και πάλι μισοψηφία απορρίπτεται. Ε, Δεύε 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρασε ψηφοφορίας. Και πάλι απορρίπτεται. Δεύε 6 υπέρ. Κατά. Ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Καταλαβαίνετε γιατί δεν υπάρχουν διαφορέ. Ξεκάθαρες, εμφανεί. Ψηφίστε παρακαλώ. Απορρίπτεται. Η ΔΕΒΕ 6, έτσι. Ναι. 97 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. 98. Θέλετε να ελέγξουμε την 96. Θέλετε να ελέγξουμε την 97. Ωραία. Ψηφίστε παρακαλώ ηλεκτρονικά για την 97. Vote is closed. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 98 υπέρ. Κατά. Ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. 98. Πέρα τη ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Με μία ψήφο διαφορά. Συμβαστική L. Υπέρ. Συμβαστική L. Υπέρ. Κατά. Ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ για τη συμβαστική L. Εκρίνεται. 103 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. 103. Three colleagues to vote. Πέρας απορρίπτεται. 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 8 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 106 υπέρ. Κατά. Ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ για την 106. Πέρα στους Εγκρίνεται 107 υπέρ κατά εποχές. Εγκρίνεται 108 υπέρ κατά εποχές. Εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία με ονομαστική κλίση. Ψηφίστε παρακαλώ. Vote is closed. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα για την εξουσιοδότηση να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. Δεν σας άκουσα. Πρέπει να ανακοινώσετε το αποτέλεσμα. 39 υπέρ 9 κατά, 6 αποχές. Νόμισα φάνηκε στην οθόνη αλλά δεν πρώτο προλάβατε. Ζητώ συγγνώμη λέει ο πρόεδρος. Ωραία. Ψηφοφορία για να δοθεί εξουσιοδότηση και να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσει με το Συμβούλιο. Όπω γνωρίζετε, με βάση τον κανονισμό χρειάζεται ειδική πλειοψηφία. Groups are thinking. Χρειάζεται ειδική πλειοψηφία, έτσι δεν είναι. Θα αφήσω λίγο λεπτά στους ε, συντονιστές των πολιτικών ομάδων να σκεφτούν την θέση τους στην τελική. Ζητώ να κάνετε λίγο υπομονή. Κοιτάξτε, για να πάει στην Ολομέλεια, ε, τεχνικά μπορώ να σας συμβουλεύσω είτε να, αναπόσχετε την ψηφοφορία να καταψηφίσετε, αν θέλετε να πάει στην Ολομέλεια. Αλλά πάντως αυτό είναι μια ψηφοφορία που πρέπει να γίνει αυτή τη στιγμή. σε κάθε περίπτωση ο εισηγητής μπορεί να εκφράσει την άποψή του, να τον ακούσουμε. Ε, θα ήθελα να επιβεβαιώσω κύριε Πρόεδρε ότι και η εισηγήτρια από τη Γιούρη και εγώ επιθυμούμε το ζήτημα να τεθεί στην Ολομέλεια. Ε, εντάξει λέει ο Πρόεδρος, ε, εκφράστε την άποψή σας, παρόλα αυτά θα κάνουμε την ψηφοφορία όπως πρέπει. Ψηφίστε παρακαλώ. Έχουμε έναν ε, υπεράριθμο ευρωβουλευτή των σοσιαλιστών. Ακόμα. Ακόμα. Συντονιστείτε παρακαλώ. Ωραία, πέρας ψηφοφορίας. Ισοψηφία, το οποίο σημαίνει ότι δεν υπάρχει πλειοψηφία, πολλό δε μάλλον ειδική πλειοψηφία, mistake of the chair, so but in... Εν πάση περιπτώσει, το μόνο σίγουρο είναι ότι θα τεθεί το ζήτημα στην Ολομέλεια. The So, is a qualified majority. Majority of. So we don't have the qualified majority. Είχα δίκιο, διευκρινίζει ο πρόεδρος. Κάτι του λέει όλος όμως από δίπλα δεν είχαμε την ειδική πλειοψηφία που χρειάζεται, είπε ο Πρόεδρος. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι η ομάδα ENF θα καταφέρει Θα υποβάλει έκθεση μειοψηφία επί του θέματο αυτού. Βεβαίω, λέει ο πρόεδρο, όπω σα είπα, θα χρειαζόταν ειδική πλειοψηφία των μελών της Επιτροπής, όχι των ε, ψηφισάντων. Έλειπαν λοιπόν πέντε ψήφοι, δεν, δεν, θα, δεν θα μπορούσε να εγκριθεί. Ε, ήθελα να το εξηγήσω. Ε, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να υπογραμμίσω, να τονίσω, ότι θα υποβάλουμε έκθεση μειοψηφίας για το, τη της αυτή, το κείμενο αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ για την ε, πληροφόρηση ε, πέρα της συνεδρίασης, ε, της κοινής συνεδρίασης με την Επιτροπή ΕΚΟΝ δηλαδή. Dear colleagues, the Committee is... Συνεχίζουμε αγαπητοί συνάδελφοι με τις εργασίες μας. Σας παρακαλούσα λοιπόν να εγκαταλείψετε την αίθουσα. Σας ευχαριστώ πολύ.